Dear colleagues, may we begin? Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε. So, welcome, welcome. Καλώς ήρθατε Καλώς ήρθατε σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών ε, Υποθέσεων. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, την ε, κυρία Ντανούτα Χούμπνερ. Να εγκρίνουμε καταρχάς την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αιτήματα για αλλαγή. Όχι. Πολύ ωραία. Οπότε θεωρούμε εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω όλους και να ευχαριστήσω τον Πάβελ ε, γιατί ε, δίνεται αυτή τη δυνατότητα προβλέποντας χρόνο για να γίνει αυτή η κοινή συνεδρίαση γιατί πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα με αυτό το θέμα. Σήμερα ε, συναντιόμαστε για να συζητήσουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης και θα ήθελα να σας πω ήδη από τώρα γιατί κάποιοι μπορεί να φύγετε. 7 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Για όσους αποχωρήσουν λοιπόν πριν από το τέλος της συζήτησης, ήθελα να το πω αυτό. Να πω επίσης ε, εισαγωγικά για ποιο λόγο είμαστε εδώ σήμερα από κοινού και οι δύο επιτροπές. Όλα ξεκίνησαν με την διοργανική συμφωνία η οποία και για τις δύο επιτροπές μας ήταν πάρα πολύ σημαντική ε, η πρόθεση ήταν να βελτιώσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τον Απρίλιο ολοκληρώσαμε ε, τη δουλειά μας για το 2016 και αποτέλεσμα αυτού ήταν ε, το Κοινοβούλιο να εντοπίσει θέματα τα οποία χρήζουν περισσότερη εργασία. Οπότε αυτό το ζήτημα το ανέλαβε μια ομάδα εργασίας ειδική ε, την οποία ελέγχουμε από κοινού με τον Πάβελ. Ήταν πάρα πολύ καλή η δουλειά. Ε, ήταν μια κοινή προσπάθεια, εξετάζουμε και ερμηνεύουμε όλα όσα έγιναν εκεί και όταν ε, ολοκληρώθηκε η εργασία της, επιτροπής ομάδας αυτής ε, τον Νοέμβριο του 2017, Προτάθηκαν, προτάθηκε μια σειρά θεμάτων να συζητηθούν. Οι δύο εισηγητέ, οι οποίοι εκπροσωπούν τι δύο επιτροπέ, ο Πάβελ Σφόμποντα και ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, μετά το πέρας ε, των εργασιών της ομάδας εργασίας ε, ολοκλήρωσαν το σχέδιο έκθεσής τους και τώρα θα τους ακούσουμε ε, και θα αποφασίσουμε πώς θα συνεχιστεί η δουλειά αυτή της έκθεσης που πιστεύω ότι θα ενταχθεί στη δουλειά και των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ντανούτα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή ε, κύριο Κόρμπετ για την εξαιρετική συνεργασία που είχα μαζί του. Είμαι βέβαιος ότι θα προσέλθει και ο κύριος Κόρμπετ ε, εντός δευτερολέπτων ή λεπτών. Η πρόοδος ε, που σημειώθηκε και η εμπειρία που αποκομίσαμε στα δύο χρόνια της διοργανικής αυτής συμφωνίας είναι σε γενικές γραμμές θετική και λογικά ενθαρρύνει τα τρία θεσμικά όργανα να προβούν σε περαιτέρω προσπάθειες να συνεργαστούν πλήρως σε σχέση με τα εκρεμή ζητήματα. Θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα ζητήματα αυτά που αναφέρει και το σχέδιο έκθεσης, γνωρίζοντας ότι δεν είχατε και πάρα πολύ χρόνο να τη μελετήσετε. Πρώτον, ε, το ιωτήσιος περιγραμματισμός ε, διοργανικός ε, υπό τη νέα συμφωνία δείχνει τη δέσμευση των τριών οργάνων και φυσικά την καλωσορίζουμε. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή ε, κατανόηση ότι η ταχύτερη ε, νομοθεσία δεν πρέπει να είναι εις βάρος της ποιότητας της νομοθεσίας. Όσον αφορά τώρα ε, τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το άρθρο 225, θα έπρεπε να ενθαρρύνεται να απαντά υπό μορφή συγκεκριμένων ανακοινώσεων που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στην παράγραφο παράγραφο 10 της νέας συμφωνίας για να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και αν η πολιτική και επίσης ε, ε, να δίνεται μια πολιτική ε, απάντηση στα πολιτικά ερωτήματα του Κοινοβουλίου. Επίσης, δικαίως η νέα συμφωνία αποσαφηνίζει ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά την πολιτική διαδικασία ούτε να δημιουργεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Η μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να καλύπτει με εξισορροπημένο τρόπο τις διάφορες πτυχές της διοργανική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 ε, μεταγραφή της ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασική ε, για την καλύτερη νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εντοπισμό του κανονιστικού υπερθεματισμού. Τα κοινοβούλια πολλές φορές έχουν αναφέρει ότι θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με διαδικασίες πριν από τη διαδικασία επιπαραβάση, ε, και στη διαδικασία επιπαραβάσης σε, επίλυση, σε μηχανισμούς επίλυσης όπως το EU Pilot που δεν θα έπρεπε να τίθεται κατά μέρο πάρα πολύ γρήγορα. Ένας τρόπος να συνεχίσουμε την διαδικασία απλοποίησης είναι μια συστηματική προσφυγή στην νομοθετική τεχνική της αναδιατύπωσης η οποία θα έπρεπε να αποτελεί την συνήθη νομοθετική τεχνική. Στην περίπτωση όμως μιας ε, ε, πλήρους ε, πολιτικής αναδιατύπωσης θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για μια εντελώς νέα πρόταση που θα ανακαλεί την υπάρχουσα νομοθεσία ώστε οι συνομοθέτες να μπορούν να δουν τα προνόμια τους να, να, να διατηρούνται όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε την πρώτη της έρευνα, ετήσια έρευνα για το φόρτο εργασίας, όπως προβλεπόταν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ε, πρέπει να γίνει μια καλύτερη επεξεργασία βάσει των ε, διδαγμάτων της πρώτης έρευνας και να εφαρμόσει μεθόδου συλλογή δεδομένων διαφανής και επαληθεύσιμους, επαληθεύσιμες, συγγνώμη, Επίσης πρέπει να τεθούν στόχοι μείωσης του φόρτου εργασίας για κάθε, καινοτομία, για κάθε πρωτοβουλία συγγνώμη, ε, βάσει ε, αξιόπιστων στοιχείων και σε πλήρη διαβούλευση με τους ε, ε ενδιαφερόμενους φορείς όπως κάνει στο πλαίσιο του Refit ήδη. Αυτά από πλευράς μου για την ώρα. Ντανούτα. Θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στο Ρίτσαρτ Κόρμπετ, αλλά δυστυχώς κάπου έχει κολλήσει μεταξύ του γραφείου του και της ε, αίθουσα. Θα του δώσουμε το λόγο πιο μετά. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση σκιωδών. Πέντε ή έξι σκιώδη εισηγητέ νομίζω είναι παρόντες ε, στην αίθουσα. Και μετά υπάρχει και κάποιος συνάδελφο άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Κάουφμαν πρώτη. Έχετε το λόγο, αν θέλετε να πάρετε το λόγο βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, λίγα πράγματα θέλω να θίξω, διότι το κείμενο της εκθέσεως μόλις χθε το έλαβα και είναι δύσκολο κατά κάποιο τρόπο να τα εξετάσω τόσο, σε τόσο σύντομο διάστημα. Πάντως, μετά από μια πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο. Είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων, όπως είπε και ο κύριος Όμποντα ο πρόεδρος μας, αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό τονίστηκε καθαρά και τονίζεται και στην έκθεση. Και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Γνωρίζουμε όλες και όλοι πόσο σημαντικές είναι αξιολογήσεις των επιπτώσεων, οι μελέτες του αντικτύπου, τα κάνει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κάνει το Scrutiny Board υπό την ιδιότητά του. Όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει αξιολογήσεις επιπτώσεων. Ίσως να μην τις κάνουμε αρκετά. Μπορούμε ωστόσο να το κάνουμε. Μπορούμε να ζητούμε από το Συμβούλιο επίσης να κάνει. Καμιά φορά ε, φοβούμε ότι πρέπει να προσέχουμε στον τομέα αυτό να μην υπερεπιβαρύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία με γραφειοκρατική ε, με γραφειοκρατία, α το πω έτσι. Μην κάνουμε δηλαδή και υπερβολικά πολλές ε, αποτιμήσεις ε, επιπτώσεων και χάνουμε κάπως το, την ευρύτερη εικόνα. Στην παράγραφο 2, μάλλον 22, διορθώνει η κυρία Κάφμαν, λέτε ότι είναι σημαντικό στις δημόσιες διαβουλεύσεις να διασφαλίζεται μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Λέτε επίση ότι δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένε ομάδε και ε, ε, μεσαίες επιχειρήσεις. Ότι αυτές είναι πολύ σημαντικές, το γνωρίζουμε όλοι, διότι είναι η σε συγκεκριμένε ομαδες πιεσεως λομπι ταυτοχρονα αυτο ραχοκοκαλιά τη επιτροπης τη εκθεσεω συγγνωμη αναφερονται παλι μικρέ και μεσαιες επιχειρήσει. οτι αυτέ ειναι πολυ σημαντικέ, το γνωριζουμε ολοι διοτι ειναι η περιφημη ραχοκοκαλια τη ευρωπαϊκή οικονομία. αλλα εαν λεμε ότι οφείλουν να ακούγονται όλες οι ομάδες συμφερόντων, να μην ε, δίνονται προτεραιότητες. Ίσως μου φαίνεται κάπως αυτό ότι δεν αρμόζει τόσο πολύ να λέγεται ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλλον, δεν, δεν πρέπει να λέγεται όταν γίνονται τόσο πολλές αναφορές στην, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το περίφημο gold plating, την επιχρήσωση των εισαγωγικών. Και αυτό το είπατε κύριε ε, Πρόεδρε. Στην έκθεση λέει, γνωρίζουμε βέβαια όταν μιλούμε για οδηγίες, γνωρίζουμε ότι οι χώρες μέλη έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να θεσπίζουν υψηλότερα πρότυπα και ότι αυτό δεν αποτελεί gold plating, για το οποίο μιλούμε βέβαια εδώ και πολύ καιρό, αλλά πρέπει να διακρίνεται διότι πρόκειται για θέματα γραφειοκρατίας από τη μια μεριά η οποία έρχεται και προστίθεται από τις χώρες μέλη μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας, αλλά η θέσπιση υψηλότερων προτύπων δεν αποτελεί gold plating. Είναι σημαντικό για τις χώρες μέλη να έχουν το περιθώριο αυτό όταν μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Ευχαριστώ πολύ. ΑΦΚΟ τώρα, ECR, ο κύριος Βιεντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Σφόμποντα για την έκθεσή του. δεν είμαι σε θέση δυστυχώς να τοποθετηθώ με λεπτομέρεια ε, επί της εκθέσεως, διότι την έλαβα μόλις χθες το βράδυ. Βέβαια, κάτι που θεωρώ σημαντικό είναι να υπάρχει ομαλή και εξορθολογισμένη νομοθετική διαδικασία που να μην επιβαρύνει υπερβολικά ιδίως τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις αλλά και τους ε, απλούς πολίτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την δική μου πολιτική ομάδα και η αδίποτε τροπολογία γίνει εκ μέρους μας αυτό το στόχο θα έχει. Την βελτίωση της προστασίας της ελευθερίας του επιχειρήν ιδίως ε, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι δηλαδή τέλο πάντων που μα. απασχολεί μας. Ευχαριστώ. ECR, Σιριάτ Καρίμ. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα ευχαριστώ τους συνεισηγητές για το στέρεο σχέδιο εκθέσεως. Υποστηρίζω πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχουν περιλάβει για τις ε, μικρές και μισές επιχειρήσεις, πρόσθετους ελέγχους αναλογικότητας και επικορικότητας, μελέτες αντικτύπων, να περιλαμβάνονται, ε, να εμπλέκονται μάλλον στην νομοθετική διαδικασία οι ομάδες ε, ενδιαφερόντων από τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας, εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν και κάποιες πτυχές που θεωρώ ότι επιδέχονται βελτίωση, για παράδειγμα η αποφυγή του gold plating. Οι σχετικές διατάξεις μπορούν να γίνουν πιο έντονες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τις προτάσεις της για μείωση του γραφειοκρατικού βάρους σε βασικούς τομείς, κάτι το οποίο θα ε, επιτρέψει σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους. Θα ήθελα να γίνουν και αλλαγές στο εγχειρίδιο μελέτης αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε το 40% των μελών να μπορούν να ζητούν impact assessments για τις τροπολογίες. Οι μελέτες αντικτύπου για τις τροπολογίες θα ενισχύσουν την θέση μας στις διαπραγματεύσεις και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ενθαρρύνονται. Το ΔΕΣ Συμβούλιο Υπουργών θα πρέπει και αυτό να ενισχύσει την εργασία του στον τομέα αυτό Κάνοντα τι δικές του μελέτες αντικτύπου με ίδρυση ειδική μονάδα. Θα ήθελα να δω και μελέτες αντικτύπου από τη μονάδα του Κοινοβουλίου, πάλι για την επικουρικότητα και αναλογικότητα, που να αναλύουν τον βαθμό κατά τον οποίο οι προτάσει, αλλά και οι τροπολογίες συμμορφώνονται με τις εν λόγω αρχές. Αυτές οι μελέτε αντικτύπου θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε ιστερότερα στάδια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο Υπουργών. Και αυτή τη στιγμή θα έχουν τροποποιηθεί σε βάθο οι προτάσει για να, να συμμορφώνονται με τι αρχέ τη επικουρικότητα και αναλογικότητα. Ευχαριστώ και πάλι του συζητητέ που λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία αυτά και αναμένω με ενδιαφέρον τι περαιτέρω συζητήσει για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ρίτσαρντ, έχετε την επιλογή. Υπάρχουν ακόμα δύο ή τρει συνάδελφοι και αν θέλετε μπορείτε μετά να μιλήσετε εσεί. Ο κύριο Καβαντά. Στο στάδιο αυτό της συζητήσεως και επειδή είναι και, και ε, πολύ σύντομε οι προθεσμίες για την ανάλυση του κειμένου, δεν θα κάνω ιδιαίτερα σχόλια. Προτιμώ να παρακολουθήσω, να ακούσω τις παρατηρήσεις των ε, παρόντων. Ευχαριστώ το έχω ακόμη τον κύριο Λεμπρετόν στον κατάλογο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εγώ επιθυμώ να τοποθετηθώ εξ ονόματος της ομάδας μου, της Ευρώπης των Εθνών και Ελευθεριών. Η έκθεση τα Κόρμπετ είναι ενδιαφέρουσα. Περιλαμβάνει πολλές συστάσεις, απόλυτα ε, καλοδεχούμενες, για την βελτίωση της νομοθεσίας για την οποία τόσο πολύ μιλούμε. Λίγες τεχνικές παρατηρήσεις, σύντομα, και μετά μια παρατήρηση πολιτική. Πρώτα, τεχνικές. Πρέπει να σέβονται περισσότερο τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Παράγραφος 4. Προθεσμίες. Εργάστηκα για την ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η οποία Γαλλική Εθνοσυνέλευση δίνει πολύ περισσότερο χρόνο για να συζητηθούν τα νομοθετήματα. Εδώ πάντοτε έχω την εντύπωση ότι πιεζόμαστε χρονικά. Το λέει και η έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα εργασιών πολύ πιο λεπτομερές και να μας το κοινοποιεί έγκαιρα για να μπορούμε να οργανωθούμε και εμείς καλύτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης οι μελέτες αντικτύπου θα πρέπει να είναι πιο σοβαρές, αυτό είναι απόλυτα ορθό αντίκτυπο ορισμένων νομοθετικών πλέον για μικρότερε και μεσαίε επιχειρήσει. Επίση, αυτή η διακρύβωση είναι πάρα πολύ ορθή. Συμφωνώ βεβαίω και με τι παρατηρήσει που έγιναν σχετικά με την αναγκαιότητα μεγαλύτερου σεβασμού και λήψη υπόψη επικορικότητα και αναλογικότητα. Από την άλλη μεριά όμω δεν συμφωνώ σε ένα άλλο πράγμα, όταν λέτε δηλαδή ότι θα πρέπει ε, να διακριβωθεί καλύτερα το κόστος της μη Ευρώπης. Μα πλάκα μου κάνετε, εάν δεν υπήρχε η Ευρώπη θα βρισκόμασταν σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον που είναι απολύτως αδιανόητο να υποθέσει κανείς ότι μπορεί να υπολογιστεί το κόστος της μη Ευρώπης. Ας σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το κόστος της μη Ευρώπης, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ας τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Και εν τέλει η έκθεση είναι καλή. Τώρα, ε, το πολιτικό σχόλιο εγώ έχω το όραμα, μαζί και με πολλούς άλλους της ομάδας μου, έχω το όραμα ενός συστήματος όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είναι ισότιμη με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, διότι από τα τρία αυτά θεσμικά όργανα ασφαλώς δύο είναι πολιτικά. Το ε, Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ή βεβαίως Υπουργών αναλόγως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει στους κόλπους του τους εκπροσώπους των λαών. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση, είναι καθαρά τεχνικό όργανο. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει μια μεταρρύθμιση που θα βάλει στη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αντικαταστήσει τον περίφημο τριμερή διάλογο με έναν διμερή διάλογο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει ένα είδο διεργού γραμματεία. Μάλιστα, Μάρκο Πίπερ. Ευχαριστώ, κυρία Ρόεδρε. Συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές για την έκθεσή τους και σε ό,τι αφορά την αναφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό, θαυμάσιο που τονίζονται τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν είναι ομάδα ενδιαφερόντων. Δεν είναι απλά ομάδα ενδιαφερόντων έχουν πολύ ξεκάθαρα αιτήματα διότι δεν έχουν τις διοικητικές ικανότητες που έχουν οι μεγάλες φύρμες. Είναι σωστό λοιπόν που διέρχεται ως ένα ερυθρό νήμα ολόκληρο το κείμενο της εκθέσεως. Το ίδιο σημαντικό είναι και το scrutiny board για τις μελέτες αντικτύπου, για τις αποτιμήσεις των επιπτώσεων. Έχουμε, πρέπει να υπερβούμε ένα κατόφλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ συμφωνώ. Για παράδειγμα, για, για τον κανονισμό της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας μιλήσαμε για το 40% χωρί καμία μελέτη αντικτύπου του Κοινοβουλίου. Τελικό συμφωνήσαμε στο 35%, πάλι όμως χωρίς μελέτη αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ορθέ μελέτε αντικτύπου. Αν όμω θέλουμε να κάνουμε και εμεί να ασκήσουμε υπεύθυνη πολιτική, πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερε αξιολογήσει των επιπτώσεων και σε άλλου τομεί τη οικονομία. Να έχουμε δυνατότητα να τι ε, διερευνούμε. Τελευταία παρατήρηση Έρχομαι σε αυτό που είπε προηγουμένω η συνάδελφό μου κυρία Κάουφμαν. Εάν οι χώρε μέλη θέτουν υψηλότερα πρότυπα από αυτά που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ίσω να μην μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό gold plating, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά όταν πρόκειται για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία των επιχειρήσεων. Είπαμε ότι υπάρχει εκεί μια εξαίρεση υπέρ των μη, μη ε, μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Ορισμένε χώρε μέλη όμω διέγραψαν ακριβώ αυτή την εξαίρεση και μέμφονται τώρα εμάς ότι αυτά όλα είναι πλέον ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εγώ όμως εδώ θέλω να μπορώ να υπερασπίσω τον εαυτό μου, να μπορώ να πω στην χώρα μου, α, μια στιγμή, αυτό σε αυτό φταίει η εθνική κυβέρνηση, η οποία κάνει αυστηρότερη την νομοθεσία από ό,τι θέλει σε το ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται αυτή η διαφάνεια. Κάθε φορά δηλαδή που οι χώρες μέλη υπερβαίνουν τα ε, ε, όσα θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να το εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες των χωρών μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ε, κυρία Χίπνερ. Θα δώσω τον λόγο στον Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Θα κάνει και εισαγωγή και τελικά σχόλια. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να φτάσω. Ο λόγο, ωστόσο ήταν λόγω ανατέρας βίας. Ευχαριστώ τον συνεισηγητή μου, κύριο Βόμποτα. Νομίζω πως έχασα μόνο την αρχική παρέμβαση, γιατί υπόλοιπα έχω κάποια γεύση των θεμάτων που αναφέρθηκαν. Εδώ βέβαια πρόκειται για την εφαρμογή των, της συμφωνίας που επετεύθη πριν από δύο χρόνια και φτιάχτηκε και αυτή η ομάδα εργασίας ανάμεσα στις ομάδες, ανάμεσα στις επιτροπές μας, όπου μπορέσαμε σε διάφορα πλαίσια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο. Ε, θέλουμε και συζητάμε να δούμε τι γίνεται. Και επίσης παρακολουθούμε τις αλλαγές στον κανονισμό Και η γενική μας εκτίμηση είναι ότι η διοργανική συμφωνία ήδη φέρνει αποτελέσματα, ήδη εφαρμόζεται και μπορεί να εκτιμηθεί θετικά. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια ε, ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. χωρίς να προσπαθούμε να ξανανοίξουμε τη συμφωνία, να διαπραγματευτούμε εκ νέου την ε, συμφωνία. Υπάρχουν ζητήματα όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα η, ε, η ε, συμφωνία. Και ορισμένα από αυτά τα θέματα είναι αυτά τα οποία θέλουμε να συζητηθούν εδώ. Καταρχήν για την επιχρήσωση δεν είναι πάντα τόσο απλό και πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στόχο έχει να εναρμονίσει ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για την ενιαία αγορά και όταν το κάνουμε αυτό θα είναι καλύτερα εκεί να χρησιμοποιούμε κανονισμούς και όχι οδηγίες για να αποφεύγουμε τις αποκλήσεις και για να ε, διατηρούμε την ομοιομορφία και εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θεσπίζει μίνιμουμ ε, προδιαγραφές και γι' αυτό και ο κύριος έχει δίκιο όταν έκανε διάκριση. Όταν ορίζουμε λοιπόν τις ελάχιστες προδιαγραφές τότε τα κράτη μέλη μπορούν να ξεπεράσουν ε, τις προδιαγραφές αυτές αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η διαφάνεια και η σαφήνεια ώστε να γνωρίζουμε πού ακριβώς το κρατημέλο, το είχε κάνει λιγότερα και πού ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει λιγότερα. Νομίζω ότι από αυτό όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ το δέχομαι ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά ότι θα πρέπει να προσέξουμε επίσης και όλους εκείνους όπου λόγω του μικρότερου τους μεγέθους ε, βρίσκονται και ακούγονται λιγότερο συχνά στις Βρυξέλλες. Οι μεγάλοι όμιλοι έχουν περισσότερες δυνατότητες να έρθουν ε, να μιλήσουν μαζί μας, ε, να παρουσιάσουν τα θέματα τους κτλ ενώ οι μικρότερες Ας πούμε υπάρχουν ομάδες ε, θυμάτων των μεγάλων φαρμακευτικών βιομηχανιών, οι ε, ομάδες καταναλωτών, οι άλλοι που ε, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν και να μας ενημερώσουν και όχι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, αυτές πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και εκείνες τις κατηγορίες όπου πρέπει να γίνουν περισσότερα και που δεν τους ακούμε τόσο συχνά. Κάτι άλλο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι μιλάμε για καλύτερη νομοθεσία και όχι για απορρίθμιση ή για κατάργηση νομοθεσίας. Οι περισσότερες νομοθεσίες ε, γίνονται για συγκεκριμένο σκοπό. Εφόσον λοιπόν νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να θυμάστε πως αυτό είναι δυνατόν εφόσον υπάρχει υψηλός βαθμός συνένεσης ότι αυτή η νομοθεσία είναι απαραίτητη. Καταρχάς χρειάζεται νομική βάση στη συνθήκη που θα ήταν αποδεκτέ από όλα τα κατημέλη όταν ενέκριναν τις συνθήκες. Δεύτερον, σημαίνει πως η πρόταση της Κομισιόν λαμβάνει υπόψη όλες τις απαιτήσει των συνθήκων σε σχέση με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα Τρίτον, χρειάζεται η έγκριση όχι μόνο αυτού του εκλεγμένου κοινοβουλίου, αλλά και του Συμβουλίου, που αποτελείται από εθνικούς υπουργούς, μέλη των εθνικών κυβερνήσεων, που είναι υπόλογοι στα εθνικά τους κοινοβούλια και χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Αυτό είναι υψηλό ποσοστό. Χρειάζεται δηλαδή υψηλό επίπεδο ε, ασφάλειας. Εκεί υπάρχει ευτυχώς ε, επαρκής έλεγχος ώστε να εξασφαλίζουμε πως η πλειοψηφία υπάρχει. Υπάρχει υψηλό επίπεδο ε, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό είναι πολύ σημαντική η ρήτρα ασφαλείας στο πολιτικό μας σύστημα. Και όσον αφορά τα σχόλια του τελευταίου ομιλητή για το ότι η Κομισιόν είναι τεχνικής φύσης σώμα, ε, ναι, η Κομισιόν δεν είναι ισότιμη με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γιατί οι νομοθέτηση είναι το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν μόνο προτείνει. Ε, Ω προ αυτό λοιπόν δεν είναι ισότιμη στην νομοθετική διαδικασία, αλλά δεν είναι ούτε και απλά τεχνικό σώμα, γιατί είναι πολιτικό, εκτελεστικό ε, σώμα, είναι υπόλογο στο κοινοβούλιο μας, εκλέγεται εδώ στο κοινοβούλιο μας και γι' αυτό ε, είναι κατά κάποιο τρόπο και πολιτικό σώμα. Ωστόσο μόνο υποβάλλει προτάσεις και το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο αποφασίζουν αν θα ε, νομοθετήσουν ή όχι και πώς. Και καλό είναι να το θυμίσουμε αυτό. Τελευταία παρατήρηση. Κάποιες φορές η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ένας τρόπος να ε, περικόπτεται η γραφειοκρατία για τις ε, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί το να έχουμε μόνο ένα σύνολο κανόνων σε μια ενιαία αγορά είναι λιγότερο περίπλοκο, λιγότερο ε, ενοχλητικό από το να έχουν 28 ε, ε, διαφορετικά σύνολα κανόνων. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στους νομοθέτες, χωρί να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει και αυτό να το υπολογίζουμε όταν εκτιμούμε κατά πόσο χρειάζεται νομοθεσία και ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσία. Δεν είναι μονόδρομος δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση αυτή. Έχουμε σημειώσει τα σχόλιά τους. Ε, έχει όμως ε, περάσει η ώρα και θα ήθελα να κάνω κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που μας περιμένει. Όπως είπα, όπως είπε μάλλον η κυρία Χούμπνερ, έχουμε μία προθεσμία τροπολογιών ε, στις 7 Φεβρουαρίου. Πρώτη εξέταση τροπολογιών θα γίνει στις 26-27 ε, Φεβρουαρίου. Μετά ε, υπάρχει μια προθεσμία για τις γνωμοδοτήσεις μέχρι τις 23 Μαρτίου και στις 26 ή 27 Μαρτίου θα υπάρξει μια δεύτερη εξέταση τροπολογιών ή ψηφοφορία. Μετά έχουμε μία χρονοθυρίδα τον Απρίλη ως ε, εφεδρική ημερομηνία και ελπίζουμε ότι θα πάει στην Ολομέλεια ή στην 1η του Μαΐου ή στη δεύτερη. Αυτά από πλευράς μου. Σας ευχαριστώ όλους ε, που ήσασταν εδώ και κυρίως την πρόεδρο ε, της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων, την κυρία Χούμπνερ. Στις 26 με 27 Φεβρουαρίου, όπως είπα, θα κάνουμε την πρώτη εξέταση ε, τροπολογιών. Συνεχίζουμε τώρα με τις εργασίες της Επιτροπής μας.